Έχετε λάβει τα εγκεκριμένα κείμενα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αντιρρήσει για τα πρακτικά. Εγκρίνονται λοιπόν τα πρακτικά ούτω. Και τώρα περνάμε.